συγκεκριμένα αιτήματα για τροποποιήσεις για τι αντιπροσωπείες και τι επιτροπέ, και θα τα δείτε στα πρακτικά. Εάν δεν υποβληθούν παρατηρήσει μέχρι την έγκριση των πρακτικών, τα ονόματα αυτά θα θεωρηθεί ότι εγκρίνονται. Στη συνέχεια